Um, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας και έχουμε την προσωρινή έκθεση της κυρίας Μακοβέη που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δίνω το λόγο για ένα τετράλεπτο στην κυρία Μακοβέη.